ή ε, μάλλον πολίτες, εκπρόσωποι του τύπου κτλ. Έχουμε λοιπόν τέσσερις κατηγορίες ψηφοφοριών με διαφορετικό βάρος, με διαφορετική βαρύτητα η κάθε μία. Παρακαλώ όσοι μπαίνουν στην αίθουσα να μην κάνω φασαρία. Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι αλλά θα είστε ακόμη πιο ευπρόσδεκτοι αν μπαίνετε ήσυχα στην αίθουσα. Έχουμε δύο κατηγορίες ψηφοφοριών που σχετίζονται με το πακέτο του προϋπολογισμού του 2011. Μετά έχουμε κάποιες μεταφορές, συνήθεις μεταφορές του προϋπολογισμού του 2010 και έχουμε και το θέμα της κυρίας Χολμάιερ για την κτηριακή πολιτική, για τα κινητά. Άσχετο θέμα, αλλά η ψηφοφορία έχει προβλεφθεί σήμερα και για το σημείο αυτό. Ως προς τον προϋπολογισμό του 2011, παρακαλώ προσοχή. Από, από το περιεχόμενο της συζήτησης ε, αντελήφθη ότι οι σοσιαλιστές, οι πράσινοι κύριε Πρόεδρε, οι φιλελεύθεροι ή γκούε. Όλες αυτές οι ομάδες ε, θέλουν αναβολή της ψηφοφορίας για τα συναφή με το ίτερ σημεία και το θέμα της ευελιξίας. Σωστά κατάλαβα. Ωραία. Καλώς. Μήπως ζητά κανείς να ψηφίσουμε για το θέμα αυτό. Γιατί αν δεν ψηφίσουμε για το σημείο αυτό, σας προτείνω να αναβάλουμε την ψηφοφορία για το θέμα αυτό σε μια έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και μάλιστα ρώτησα ποιες είναι οι ελεύθερες ημερομηνίε. Θα σας στείλουμε φυσικά και γραπτή πρόσκληση, επιβεβαίωση μάλλον. μπορούμε να συνεδριάσουμε τη Δευτέρα 13 ε, Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο 9.30 με 10.30 το βράδυ στην αίθουσα WIC 100. Αυτή είναι η δυνατότητα ο πρόεδρος των Πρασίνων. Αν κατάλαβα καλά, εμείς ζητήσαμε αναβολή για του χρόνου, όχι για τώρα, όχι για την άλλη εβδομάδα δεν θέλουμε να ψηφίσουμε σήμερα, αλλά ούτε και την επόμενη εβδομάδα, 13 Δεκεμβρίου. Να ψηφίσουμε λοιπόν ως προς την αναβολή της ψηφοφορίας έκθεσης Μπέγκε και των συναφών θεμάτων για την επόμενη χρόνια. Ε, μπορεί να είναι παράδοξο, αλλά έτσι έχει ζωή. Κύριε Καρίγκα, σε λίγο θα σας δώσω το λόγο αν επιμένετε. Ως πρόεδρος έχω τη δυνατότητα να αποφασίσω για το περιεχόμενο της σημερινής διάταξης. Διαπιστώνω λοιπόν ότι πολλές ομάδες δεν θέλουν να ψηφίσουμε σήμερα. Αποφασίζω λοιπόν ότι δεν θα ψηφίσουμε σήμερα για το σημείο αυτό. Και θα δούμε τη Δευτέρα, εντάξει. Συμφωνείτε του τέστην. Θα προσπαθήσω να διασφαλίσω για όσο μεγαλύτερο διάστημα γίνεται την ενότητα και τη σύμπνοια στους κόλπους της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και ευχαριστώ όσους θα με βοηθήσουν σε αυτό το έργο. Και ευχαριστώ και τους υπόλοιπους που θα μου δώσουν την ευκαιρία να φτάσω σε κατάσταση νιρβάνα Το πλεονέκτημα αυτής της κατάστασης είναι ότι τρεις ψηφοφορίες αναβάλλονται. Και το θέμα αυτό θα μας απασχολήσει και πάλι τη Δευτέρα. Θα ήθελα να επισημάνω και για το κοινό που μας παρακολουθεί και για τους εκπροσώπους των άλλων θεσμικών οργάνων ότι στο μεταξύ θα λάβει χώρα και ένα Συμβουλίο Υπουργών που θα αποφανθεί ως προς τις προτάσεις της ΚΟΡΕΠΕΡ για το θέμα αυτό θα συνεδριάσει αύριο το πρωί η διάσκεψη των Προέδρων των ομάδων που θα επιληφθεί του θέματος και θα αποφασίσει για το τι μέλη γενέστε και ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα εξέτασης των διάφορων πτυχών του δημοσιονομικού πακέτου για την Ολομέλεια. Η Επιτροπή Προπολογισμού θα ξανασυνεδριάσει τη Δευτέρα και η διάσκεψη των Προέδρων θα αποφασίσει αν θα μπει στην Ολομέλεια το θέμα αυτό, είτε την επόμενη εβδομάδα, είτε του χρόνου όπως προτείνουν μερικοί, είτε το 2012. Άρα, το σημείο για την ευελιξία, το 2-1. Το 2-2 για το σχέδιο έκθεσης Ράιμερ Μπέγκε, για τη διοργανική συμφωνία που αφορά το ΙΤΕΡ. Το σημείο 2-3 διορθωτικό προπολογισμό του 2010. Αυτά τα τρία συναφή θέματα αναβάλλονται. Οπότε, ο Ράιμερ διαδικαστικό. Με, πά, με όλο το σεβασμό κύριε Πρόεδρε, το πακέτο αυτό δεν έχει πλέον το όνομά μου, δεν φέρει πλέον το όνομά μου. και θεωρώ ότι η απόφαση για το κατά πόσο το ίτερ ή το μέσο το ευελιξίας θα πρέπει να αναβληθεί όχι είναι αρμοδιότητα της διασκέψης των Προέδρων. Δεν θα έπρεπε να αναλάβουμε τέτοια ευθύνη. Δεύτερη παρατήρηση. Σημειώνω ότι εδώ στην Επιτροπή μας αλλά και σε όλο το Κοινοβούλιο δημιουργείται η εντύπωση σαν ο για να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα του Κοινοβουλίου έχει ταχθεί τουλάχιστον ε, για τη διατήρηση των μηχανισμών ευελεξίας και ε, αναφέρθηκε ότι πολέμησε γι' αυτό και μετά άφησε τους υπόλοιπους συναδέλφους ε, στα κρύα του λετρού αρνούμε αυτή την κατηγορία με πάσα σαφήνεια ότι πουλάω τα συμφέροντα του Κοινοβουλίου. Και διαφωνώ, με την πλειοψηφία προφανώς της ε, Επιτροπής για το πότε θα πρέπει να ψηφιστεί αυτή, αυτός ο συμβασμός με το Συμβούλιο. Και γι' αυτό παρακαλώ αυτές τις δύο εκθέσεις και για την προσαρμογή του κανονισμού του δημοσιονομικού πλησίου. Ζητάω λοιπόν να με απαλλάξετε από την υπευθυνότητα, από την αρμοδιότητα για τη σύνταξη αυτών των εκθέσεων και μέχρι τότε θα πρέπει εσείς κύριε Πρόεδρε να λάβετε και να είστε ο εισηγητής για τις δύο αυτές εκθέσεις και πραγματικά δεν βλέπω άλλο τρόπο παρά να ακολουθήσω τον δρόμο αυτό που προτείνω. Euh. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Ράιμαρ. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε την ψυχική σας κατάσταση και νομίζω ότι όλοι υποκλεινόμαστε μπροστά στις ε, ικανότητές σας και στην αξιοπρέπειά σας και νομίζω ότι ελπίζω αν κάτι ακούστηκε στραβά μάλλον έγινε παρερμηνία ήταν με ένας παραλυσμός ε, με τη βίβλο ε, λάθος ήταν ε, παρερμηνία έγινε χαίρομαι που είστε μαζί μας και ήταν τιμή για μένα που ήμουν ο δικός σας διάδοχος και θα σας διαδεχθώ και στην έκθεσή σας θα αναλάβω εγώ την έκθεση από εδώ και πέρα. Ο κύριος Γκαρίγκα θέλει τίποτα για την διαδικασία των ψηφοφοριών, όχι αργότερα. Καλώς. Στρέφομαι τώρα προς τους συγγητές. Θα χρειαστείτε και τις ηλεκτρονικές κάρτες ψηφοφορίας. Αχρίαστες να είναι, αλλά δεν βλέπω και πολύ μεγάλη ομοφωνία σήμερα το απόγευμα και απόλυτη σύμπνοια, οπότε ας έχουμε για καλό και για κακό τις ηλεκτρονικές κάρτες ψηφοφορίας. Τον φρονίμα τα παιδιά. Λοιπόν, κυρία εισηγητρία, πώς προτείνετε να διοργανώσουμε τις ψηφοφορίες για τον προϋπολογισμό του 2011. Υπάρχει πλειοψηφία, όχι ομοφωνία, αλλά υπάρχει πλειοψηφία να ψηφίσουμε με βάση αυτά που προτάθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τροποποιήθηκαν από την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων. Για τεχνικούς λόγους όμως θα χρειαστεί να ψηφίσουμε... Θα μπλοκαριστούν πολλά σημεία, θα χρειαστεί να ψηφίσουμε διάφορες τροπολογίες. Κυρία εισηγητρία, εσείς καταρχήν πώς θέλετε να προβούμε στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι σημαντικό να πούμε κάτι που είναι σαφές για τους ε, περισσότερους, αλλά όχι για όλους, ότι πρόκειται για ένα κοινό εγχείρημα μεταξύ μου και της Χέλγκα Τρούπελ. Και για το τρίτο τμήμα, αλλά και για άλλα τμήματα. Η ψηφοφορία, λοιπόν, όχι ότι είμαστε δύο άτομα και πρέπει να μας κατηγορείτε, αλλά τέλος πάντων είναι σημαντικό να το δούμε αυτό σε ενότητα. Η ιδέα του να ψηφίσουμε, όπως σας εξήγησα και σε ένα email που σας έστειλα, η ιδέα είναι λοιπόν να ψηφίσουμε πρώτο για τα ποσά και για τις παρατηρήσεις, τρίτο τμήμα και άλλα τμήματα, μετά να ψηφίσουμε για τα αποθεματικά και τρίτο τμήμα και άλλα τμήματα και τέλος για τον πίνακα που, ψηφι... που συζητήσαμε και προηγουμένως. Μεταξύ των ψηφοφοριών αυτών να γίνει και ε, ψηφοφορία για τις τροπολογίες για τους ίδιους πόρους. Δύο τεχνικές παρατηρήσεις έχω να κάνω ανακοινώσεις. Επειδή ανακαλύψαμε ότι κάποιες από τις παρατηρήσεις επί των οποίων είχαμε συμφωνήσει για κάποιους τεχνικούς λόγους δεν παρουσιάστηκαν στη νέα, στο νέο σχέδιο προπολογισμού που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά έχουμε συμφωνήσει ότι θα ενσωματωθούν. Αυτό στην πράξη τι σημαίνει ότι στη σειρά διορθώθηκε μια τέτοια παρατήρηση από τη Χέλικα Τρούπελ. Άρα εδώ είναι ένα ζήτημα που θα ήθελα να υπερψηφίσουμε. Πρόκειται για την τροποποίηση 003 στο 080401 και κάτι άλλο σε ό,τι αφορά την γραμμή για την γραμμή 150555 για το πρόγραμμα Youth in Action, νεολαία ενδράση θα ήθελα να συμπεριληφθεί και ως προφορική τροπολογία, αλλά έχει, ε, το έχουμε ήδη συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει παραληφθεί απλά για τεχνικούς λόγους. Αυτά από δική μου πλευρά. Για τις τροπολογίες για τα ποσά, δεν θα σας προκαλέσει έκπληξη και για τις να αναφέρω ότι πέρα από την τροπολογία που επανακατέθεσε η Χέλγκα Τρούπελ, θα ήθελα να σας συστήσω να τις καταψηφίσετε όλες. Θα μπορούσαμε ενδεχομένω να τις ψηφίσουμε ε, όλες μαζί αν μπλοκ. Αυτό θα μας διευκόλυνε. Αν όχι, μπορούμε να τις ψηφίσουμε και μία προς μία. Για τα αποθεματικά, δεν νομίζω ότι μπορούμε να ψηφίσουμε συνολικά γιατί όπως σας είπα έχουμε 8 συν 3 αποθεματικά. Θα ήθελα να ψηφίσουμε υπέρ 5 αποθεματικών, άρα θα πρέπει να γίνει ξεχωριστή ψηφοφορία. Αυτά από πλευρά μου. Bien. Καλώς. Η πρώτη ψηφοφορία αφορά την ενεργοποίηση του μέσου ευελιξίας. Δεν έχει καμία σχέση με την προηγούμενη συζήτηση. Είναι συνώνυμα απλώς είναι μάλλον ταυτόσιμε έννοιε. Είναι μια δημοσιονομική γραμμή που μα επιτρέπουν υπέρβαση των ανώτερων ορίων και θα πρέπει να ψηφίσουμε ξεχωριστά για το μέσο ευελιξία. Η συγκεκριτή για το θέμα αυτό ήταν ο Ράιμερ Μπέγκε, τον διαδέχομαι εγώ, 500 εκατομμύρια. Η ενεργοποίηση αυτού του μέσου ευελιξία θα μα επιτρέψει να χρηματοδοτήσουμε όλες τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για πιστώσεις ανάληψη υποχρεώσεων για το 2011. Ποιος είναι υπέρ? Υπέρ. Ωραία. Κατά. Δύο ψήφοι κατά. Αποχές. Μεγάλη πλειοψηφία. Δεν χρειάζεται καν ηλεκτρονικός έλεγχος. Ωραία. Περνάμε στον πίνακα, τον κατάλογο της ψηφοφορίας. Τρίτο τμήμα. Έχετε όλοι τον κατάλογο, μπορείτε να ψηφίσετε. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω και φυσικά θα ψηφίσουμε ξεχωριστά τις τροπολογίες. Αν τελικά σε επίπεδο ολομέλειας, σε επίπεδο ε, Συμβουλίου, Υπουργών στο Συμβούλιο και Ολομέλεια στο Κοινοβούλιο, αν δεν έχουμε παρόμοια ψήφο σε όλες τις γραμμές, θα χρειαστούμε συνδιαλλαγή. Οπότε, για το 2011, για τον προπολογισμό αυτό, στόχος μας είναι το συντομότερο δυνατό να, φτάσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία και αντίστοιχη ψηφοφορία. Ομοιότητα στη στις ψήφους. Θα υπάρξουν κάποιες διαφωνίες, ιδιαίτερα για τα αποθεματικά από ό,τι φαίνεται. Για την κατηγορία 1α έχουμε την τροπολογία 18 του κυρίου Ζόντερκαρτ της Γκουε. Η συγκέντρια είναι κατά ποιος είναι υπέρ. Κατά. Τέσσερις ψήφοι υπέρ, οι υπόλοιποι κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12, Goran Firm. Η συγκέντρη είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Η πλειοψηφία είναι κατά. Δύο αποχές. Απορρίπτω ο κύριος Πόρτας ζήτησε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αν θέλετε να διευκολύνετε τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Οι τροπολογίες της ΓΚΟΕ να ψηφιστούν μπλοκ, ανακεφάλαιο, όχι ξεχωριστά. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αν και άλλοι μιμηθούν το παράδειγμά σας, θα είμαστε ευγνώμονες. Προτείνω λοιπόν, μετά την πρόταση του κ. Πόρτας, τις τροπολογίες 38 έως 22, 41, 39, 40, 42, 43, 17 και 22 καθώς και την τροπολογία 21, που είναι όλες οι τροπολογίες της ΓΚΟΕ, στην κατηγορία 1α, να τις ψηφίσουμε, ανα, ανακατηγορία θα ψηφίσουμε, να τις ψηφίσουμε όλες μαζί. Ο κύριος Πόρτα συμφωνεί, η εισηγήτρια είναι κατά, ποιος είναι υπέρ. Ο κύριος Πόρτας, κατά. Πολύ και διάφοροι. Αποχές, ωραία. Κύριε Πόρτας, Μόνο εσείς είστε, δυστυχώς δεν έχετε πλειοψηφία. Απορρίπτονται όλες οι τροπολογίες αυτές που αναφέραμε. Τροπολογία 49 τη κυρία Αντρέασεν. Η συγκίτρια είναι κατά. Ποιο είναι υπέρ. Δύο υπέρ. Κατά. Η πλειοψηφία. Αποχές. Μία αποχή. Απορρίπτεται και αυτή. Τροπολογία 3 της κυρίας Τρίπελ. Η συγκίτρια είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Τέσσερις. Αποχές μία αποχή, εγκρίνεται. Τροπολογία 50, Ανδρέασεν. Η συγκέντρη είναι κατά. Ποιο είναι υπέρ. Η κυρία Ανδρέασεν φαντάζομαι είναι υπέρ και άλλοι δύο. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 1, Έλγα Τρίπελ. Η συγκέντρη είναι κατά. Εδώ ποιο είναι υπέρ. Η πράσινη είναι υπέρ. Και ο κύριος Πόρτας. Κατά, πολύ είναι κατά. Αποχές. Μία αποχή. Η Αν Γένσεν ζητάει το λόγο για διαδικαστικό. Με ενέπνευσε το παράδειγμα του κυρίου Πόρτα. Γι' αυτό θα έλεγα να ψηφίσουμε μαζί όλες τις τροπολογίες της Φιώνας Χολ που είναι ομοειδεάτησα. Καλώς. Σας ευχαριστώ για το πνεύμα συνεργασίες που δείχνει η Αν Γένσεν. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Το περιμένουμε από εκείνη. Ωραία, ψηφίζουμε όλε τι τροπολογίε τη κυρία Φιώνα Χολ για την κατηγορία 1α, γιατί ψηφίζουμε ένα κατηγορία. Δηλαδή, λοιπόν, τροπολογιε 009 ως 005. Η συγκέντρη είναι κατά, ποιο είναι υπέρ. Τροπολογία 04 ως 09, 05, συγγνώμη. υπάρχει διάσταση απόψεων, διβυσιών ταπεινιώνες όπω λέμε στα ισπανικά, λέει ο πρόεδρο ηλεκτρονική επαλήθευση. Οι τροπολογίε 04, 09, 08, 07, 06 και 05. Τροπολογίε τη κυρία Φιώνα Χολ. Απ, περισσεύει ένας σοσιαλιστή. Και από το ΕΛΚ επίση. αλλά για το ΕΛΚ είναι εύκολο, όπως ήρωμαι εγώ. Σοσιαλιστέ. η Γιούτα, εντάξει. Η Γιούτα και εγώ δεν θα ψηφίσουμε. Βγάζω την κάρτα μου από το μηχάνημα. Ψηφίζουμε τις τροπολογίες Φιώνα Χολ. Η συγκέντρια είναι κατά. Άρχεται η ψηφοφορία. Γιούτρα, Γιούτα μην ψηφίζεις. Άρχεται η ψηφοφορία. Ίγκε ψήφισε. Τέλος. Αποτέλεσμα. 19 pour 22 contre. 22 η 19 υπέρ 22 κατά το αντίστροφο είπε ο πρόεδρος έχουμε δύο τροπολογίες της ΓΚΟΕ η συγκεκριμένη είναι κατά ποιος είναι υπέρ μόνο ΓΚΟΕ κατά όλοι οι υπόλοιποι αποχές χωρίς αποχές κύριε Πόρτας πάλι μόνο σας είστε απορρίπτονται οι τροπολογίες σας Περνάμε στη δεύτερη κατηγορία, μια σειρά από τροπολογίε του κυρίου Χάουζερ που δεν είναι εδώ. Λοιπόν, άντε, θα τι ψηφίσουμε αν μπλοκ. Η συγκίτρια είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Τι είναι εδώ, ο κύριος Σερενάουζερ. Α, με συγχωρείτε. Ναι, συγγνώμη. Φυσικά και είμαι εδώ και δεν θα ήθελα να ψηφίσουμε αν μπλοκ. Ναι, με ακούτε. Τέλεια. Ναι, εννοείται ότι είμαι εδώ και δεν ζήτησα να ψηφίσουμε blog. Θα ήθελα να τις ψηφίσουμε ξεχωριστά. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Δεν ε, είχα δει ότι ήσασταν εδώ. Ε, τώρα που διαπιστώνω πως είστε παρόν, δέχεστε να ψηφίσουμε ένα ναι, αυτό ήθελα να πω ότι όχι, δεν συμφωνώ. Wow. Δικαίωμά σας. Δικαίωμά σας. Οι συνάδελφοι θα το εκτιμήσουν όλο ιδιαίτερο. L'amendement 57, qui est Τροπολογία 57, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 66 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έχουμε μία τροπολογία της Γκουε όχι έχουμε διάφορες της Γκουε λοιπόν 19, 20, 44, 45, 46, 47, 48. Αυτά για την κατηγορία H1Β με την ευγενική συμφωνία του κυρίου Πόρτας τις ψηφίζουμε σε unblock. Ε, Ποιοι είναι υπέρ, η είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ, κύριος Πόρτας είναι βεβαίως υπέρ. Ποιοι είναι κατά, δυστυχώς η μεγάλη πλειοψηφία. Άρα απορρίπτονται. Ερχόμαστε στην 68 του κυρίου Έραν Άουζερ. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 69, το ίδιο συντάκτη. Η συγκεκριμένη είναι κατά, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 70 του κυρίου Έραν Άουζερ, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Επιστώνω ότι ο κύριος Έραν δεν υπερψηφίζει τις τροπολογίες του, αλλά εν πάση περιπτώσει ψηφίζουμε. Μετά πάμε στην 71. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Στη συνέχεια έχουμε όλες τις τροπολογίες της Γκουε και... Α, ναι, ωραία, τελειώσαμε με την ε, ε κατηγορία 2. Πάμε στην 3α, κατηγορία 3α. Έχουμε την, εισηγής, την ε, τροπολογία Αντρέασεν, η εισηγή την κατά, ποιοι είναι υπέρ, η κυρία Αντρέασεν, 1, 2, 3, 4. Και ο κύριος Στάς, μάλιστα. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έχουμε στη συνέχεια μια μεμονωμένη τροπολογία της ΓΚΟΕ, την 24. Η εισηγήτρια είναι κατά, υπέρ, 3. Κατά αποχές απορρίπτεται. Μια μόνο τροπολογία στην κατηγορία 3β που είναι πάλι της ΓΚΟΕ, η συγκεκριμένη κατά, ποιοι είναι υπέρ. Τέσσερις. Αυξάνονται κατά αποχές απορρίπτεται. Κατηγορία 4. Έχουμε μια σειρά από τροπολογίες της ΓΚΟΕ που αντιστοιχούν σε τρεις τροπολογίες που είναι κάτω-κάτω και γυρνάω τη σελίδα, μετά έχω τις τροπολογίες 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 και 35. Ο εισηγήτρια είναι κατά, ψηφίζουμε αν μπλοκ, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Πάμε στην 76 της κυρίας Αντρέασεν. Η συγγήτρη είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Φτάνουμε σε μια άλλη τροπολογία της κυρίας Αντρέασεν, την 68. Ο εισηγητής είναι 78, συγγνώμη. Ε, ε, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ακολουθεί η τροπολογία 2 για την μπανάνα της κυρίας Τρούπελ. Η συγκεντρία είναι κατά, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Πλειοψηφία είναι κατά. Πράσινοι και οι σοσιαλιστές είναι μια ψηφία για την μπανάνα. Απορρίπτεται. Euh, alors, nous passons Κατηγορία 5. Τρεις τροπολογίες του κ. Ερενχάουζερ. 80. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 81. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Μία. 83. Υπέρ. Κατά. Κατά. Αποχές. Μία αποχή απορρίπτεται. Για τα υπόλοιπα τμήματα. Έχουμε την τροπολογία 87 της κυρίας Ανδρέασεν. Η είναι κατά, ποιον υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 90. Ερενάουζερ, η συγγήτρια είναι κατά, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Ευχαριστώ αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία πολύ αγαπημένη για τους ίδιους πόρους. Αλλά η συγγήτρια είναι κατά, ποιοι είναι υπέρ, κατά. Η ίδια πλειοψηφία όπως πριν. Αποχές και δεν μπορώ και να ψηφίσω γιατί είναι πολύ από το ΕΛΚΑ εδώ. Ελπίζω. Ελπίζω πως ο πρόεδρος της ομάδας των Πρασίνων θα μετρήσει, θα καταλάβει το μαρτύριο το οποίο περνώ. Ναι, ναι, είναι αλήθεια. Ναι, θα χρειαστώ λίγες μέρες ε, λιγότερο κάθαρση. Και έπειτα τον, ε, τον αντιμετωπίζω τον ε, πρόεδρο των Πρασίνων θα μου κοστίσει και παραπάνω. Λοιπόν, τροπολογία 14, Γκόραν Φέρμα, υπέρ κατά ίδια πλειοψηφία, αποχές, απορρίπτεται. Alors, sur les nouvelles, nouvelles autorités. Alors, nous passons maintenant au vote des amendements sur les réserves. Alors là... Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία για τα αποθεματικά. Εδώ λοιπόν, και μιλώ υπό τον έλεγχο της εισηγητρίας, εδώ προτείνω unblock πάλι τροπολογίες για να είμαστε συνεπείς για ό,τι αφορά την κατηγορία 1α πρόκειται για επιφυλάξεις, ε, για αποθεματικά με για τους νέους οργανισμούς. Όλα τα αποθεματικά λοιπόν της κατηγορίας 1α, η συγκήτρια είναι υπέρ, ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Ένας μια Μία. Τώρα. 3α. Το ίδιο. Unblock. Όχι, όχι. Γιατί είναι δύο διαφορετικές αρχές. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε το sis 2. Πριν από λίγο, ο Γενικός Διευθυντής εξέφρασε μια ανησυχία για ένα αποθυματικό 100%. Αυτή η ανησυχία οδηγεί την εισηγήτρια να αλλάξει την πρότασή τη Πείτε μου ναι ή όχι απλώς και απλώς θα ψηφίσουμε. Όχι. Ωραία, ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε την τροπολογία 72. Ποια είναι υπέρ. Κατά. Ένας. Αποχές. Υιοθετείτε. 73 για την Ευρωπαϊκή ε, Αστυνομική Ακαδημία. Το Συμβούλιο την θέλει πολύ αυτή. Πιπέρ, κατά. Αποχές. Μία. Εγκρίνεται. Τώρα έχουμε την κατηγορία 3β. Η συγγήτρια είναι αντίθετη. Δηλαδή αποσύρεται. Αποσύρεται. Μάλιστα. Είναι πιο απλό. Ε, τώρα, ε, πάμε στην κατηγορία 4. Τροπολογία 77. Ναι, με συγχωρείτε. Ναι, εισηγήτρια, έχω ένα σχόλιο. Εγώ διστάζω να τις αποσύρω αλλά, γιατί τις ε, ως εισηγήτρια αλλά δεν τις έχω συντάξει εγώ. Είναι τροπολογίες που έχουν επανεποβληθεί και γι' αυτό και προτείνω να ψηφιστούν παρότι εγώ είμαι αντίθετη. Έφτασαν νέες πληροφορίες και έχω αλλάξει την άποψή μου για το αποθεματικό αλλά μπορεί να υπάρχουν κάποιοι που να διαφωνούν μαζί μου και να έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν. Eh, Μια στιγμή. Θέλετε να ψηφίσουμε την 75? Εντάξει, εντάξει. 75. Η συγκέντρη είναι κατά γιατί άλλαξε γνώμη. Ποιο είναι υπέρ. Κανεί. Κατά. Όλοι. Ε, Κανεί δεν είναι υπέρ, ήταν σαν να δεν είχαμε αποσύρει. 77 τη συγκεντρία. Ποιο είναι υπέρ κατά απο, αποχές, δύο ψήφοι κατά, χωρίς αποχές, εγκρίνεται. 11 του Γκέραν Φέρμ. Η εισηγήτρια είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Η αριστερά. Κατά. Η δεξιά και το κέντρο. Αποχές. Η ίδια, η ίδια πλειοψηφία προηγουμένως για την μπανάνα. Φαίνεται ότι ο Γκόρεν Φέρμ πήρε τη σκητάλη από το Λάζο Σούριαν που αποουσιάζει για τι μπανάνε. Κατηγορία 5. Τροπολογία 79. ποιο είναι υπέρ. Κατά. Μία ψηφο, κατά αποχέ. Χωρίς αποχέ. Εγκρίνεται. 10. Τον Γκόρεν Φέρμ. Η συγκέντρια είναι κατά. Ποιο είναι υπέρ. υπάρχουν πιο πολλέ ψήφοι υπέρ. ηλεκτρονική επαλήθευση ούτε εγώ ψηφίζω ούτε η Γιούτα. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Τέλος. 21-21. Ισοπαλία. Άρα απορρίπτεται η τροπολογία. 82. Δύο τροπολογίες. Είναι για δύο δημοσιονομικές γραμμές. Η Σιδόνια δεν αποσύρει τροπολογία της. θα ψηφίσουμε μία φορά τα δύο σκέλη της 82. Η σύγκριτρια είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Η πλειοψηφία είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτονται τα δύο σκέλη της 82. 84 για τους ειδικούς συμβούλους. Η σύγκριτρια είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Μερικοί ψήφισαν και υπέρ και κατά. Τι θα πει αυτό. Μάλλον κατά. Καλά, ηλεκτρονικός. Η Σκανδιναβοί δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Γιατί ξέρουν στον παγετό πόσο να οδηγούν. Για να γυρίσει κανείς φαίνεται να κάνει τετακέ. Για το 85 η συγκέντρη είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ κατά, δύο κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 86, Ερενχάουζερ. Η συγκέντρια είναι κατά, ποιος είναι υπέρ. Κατά, ευχαριστώ, αποχές, απορρίπτεται. Λοιπά τμήματα για τα αποθεματικά και πάλι. Δύο τροπολογίες, έλεγα Τρούπερ, να τις ψηφίσουμε μαζί, κυρία Συγκέντρια Συγγνώμη, δε, είναι η προπολογισμό τη Χέλγα, δεν είναι τη Συντόνια πια. Αντικαθιστά κάποιο την Χέλγα. Μαζί τι τροπολογίε, η γιατρή είναι υπέρ των δύο τροπολογιών. Ποιο είναι υπέρ, 88 και 89. Κατά. Αποχέ, μία ψήφο κατά, χωρί αποχέ εγκρίνονται. Ψηφίζουμε τις 15 και 16 του Γκέραν Φέρ μαζί. Ποιος είναι υπέρ, Κατά. Δεν συγκεντρώνεται πλειοψηφία, άρα απορρίπτονται παρά την υποστήριξη της ηγετριάς. Ψηφίζουμε τώρα το σύνολο των πινάκων που αφορά, αφορά την επιχείρηση μισθή. Και για να απαντήσω στην ερώτηση που έθεσε πριν στη Χέλκα Τρίπελ, η οποία μα εγκατέλειψε προ στιγμή, η χρηματοδότηση τη επιχείρηση μισθή δεν θα έχει αρνητικέ συνέπειε, αρνητικό αντίκτυπο στον στο λειτουργικό προπολογισμό των θεσμικών οργάνων και μάλιστα θα έχει και θετικέ συνέπειε. Γιατί κατ' εκτέλεση τη νομολογία του ΔΕΚ θα έχουμε αύξηση των μισθών, θα είναι θετική συνέπεια, αλλά αρνητικέ συνέπειε δεν υπάρχουν. Οπότε φαντάζομαι ότι η συγγέντρια για τα λοιπά τμήματα είναι υπέρ. Ψηφίζουμε λοιπόν τους πίνακες μαζί. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Δύο. Αποχές. Μία αποχή. Σας ευχαριστώ. Οπότε ολοκληρώνουμε για τα ποσά. Έχουμε το ψήφισμα τώρα. Οι συγητές υποβάλλουν στην Επιτροπή Προϋπολογισμών ένα ψήφισμα που θα το χαρακτήριζα αμυγός περιγραφικό. as supported by the Green Rapporteur. But Sedonia was again. Sur, sur la déclaration, donc. Για τη δήλωση. Κανονικά είναι, έχει περιγραφικό χαρακτήρα, αλλά υπάρχουν και τροπολογίες. Οι συντάκτες είναι πολλοί. Καταρχήν, τροπολογία εναρτών. γιατί είναι κατά ποιος είναι υπέρ. Κύριο Αρτόγκ φυσικά είναι υπέρ. Δύο υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Κατόπιν έχουμε τρει ε, τροπολογίε ε, του κυρίου Χάγκλουντ. Ερωτώ του φιλελευθέρου αν μπορούμε να τι ψηφίσουμε μαζί. Όχι. Καλά. Τροπολογία 2. Άγκλουντ. Η συγκίτρια είναι κατά. Ποιο είναι υπέρ. Ωραία. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος, παρακαλώ. Η Γιούτα και εγώ δεν ψηφίζουμε. Τροπολογία 2, άρχεται η ψηφοφορία. Σασπένς, 19 υπέρ, 21 κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3, Χάγκλουντ. Η συγκέντρια είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Και εποχές ε, οι σοσιαλιστές απέχουν. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4 Χάγκλουντ. Η συγκίτρια είναι κατά ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία και νομίζω ότι είναι η ίδια πλειοψηφία. Αλλά στο ελέγξουμε καλύτερα. Γιατί είναι περίεργες αυτές οι πολιτικές συμμαχίες. Ασυνήθιστες. Μας έχει μπερδέψει ο κύριος Χάγκλουντ. Τέλος ψηφοφορίας για την τροπολογία 4, 19 υπέρ 23 κατά, ίδια πλειοψηφία με προηγουμένως, απορρίπτεται. Τροπολογία 5 του κυρίου Χάρτονγκ. Ποιος είναι υπέρ. 2 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Νέα τροπολογία Χάγκλουντ, υπαριθμόν 6. Η συγκέντρια είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. επανάληψη ψηφοφορίας με ηλεκτρονικό τρόπο γιατί έχω την αίσθηση ότι έγινε κάποια μικρή αλλαγή στις συμμαχίες. Ψηφίσατε όλοι, τέλος ψηφοφορίας για την τροπολογία 6. 19 υπέρ, 20 κατά, 2 αποχές. Όντω μια μικρή αλλαγή έγινε, αλλά παρόλα αυτά απορρίπτεται και πάλι η τροπολογία. Τροπολογία 7 αγγλούν και 8 Αχτών, πανομοιότυπες. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 7 και 8. Τέλος ψηφοφορίας. 20 υπέρ, 21 κατά. Οριακή διαφορά, αλλά απορρίπτονται οι δύο τροπολογίες. Ψηφίζουμε την έκθεση. Ονομαστική ψηφοφορία, ηλεκτρονικά, τελική ψηφοφορία για το ψήφισμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 27 υπέρ, 5 κατά και 10 αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν. Συγχαρητήρια κυρία εισηγητρία. Μπράβο σας. Και ευχαριστώ και τα μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών. και συγχαρητήρια και στην Έλγα Τρίπελ. Σα ευχαριστώ όλου για τη συνεργασία σα. Α, δεν τελειώσαμε, δεν τελειώσαμε. Ο κύριο Άλβαρο θέλει το λόγο. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ήθελα να παρέμβω. Αφού έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας έναν εκπρόσωπο της διάσκεψης των Προέδρων που έχει αυτό το, δεύτερο, το διπλό καθήκον. Είναι μέλος της Επιτροπής μας και μέλος της διάσκεψης των Προέδρων. Αυτό που έλεγε και είπε προηγουμένως ο συνάδελφος Μπέγκη είπε ότι θέλει να αποσυρθεί το όνομά του από την έκθεση. Αυτό δεν ελήφθη υπόψη. Εγώ γνωρίζω τον κύριο Μπέγκε εδώ και έξι χρόνια και Πραγματικά δεν το έχω δει να επαναλαμβάνεται αυτό. Μόνο όταν υπάρχουν αντιρρήσει για θέμα περιεχομένου ή για διαδικαστικά θέματα τα οποία δεν ε, βρίσκουν σύμφωνο τον εισηγητή. Γι' αυτό το λόγο και η δική σας ε, στη συμμετοχή εδώ ε, ήταν πολύ σημαντική όσον αφορά τα διαδικαστικά θέματα. Θα έχουμε ολοκληρώσει, παρακαλώ, να στρέφουμε στους συντονιστές της Επιτροπής ε, Προϋπολογισμού να λάβουν υπόψη το θέμα με τη... και με τους ε, προέδρους να δουν ακριβώς το θέμα των αρμοδιοτήτων. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αρμοδιότητα αυτής της Επιτροπής που θέλουμε να απλοποιήσουμε δηλαδή μια παλιά συνήθεια της διάσκεψης των Πρόεδρων. Όχι. Και γι' αυτό έχουμε και για τον κανονισμό μαζί μας. Ναι, αλλά ξέρετε ότι πρέπει και αυτό να το ακούσετε. Δεν είναι δυνατόν. Μπορούμε να μιλάμε στην Ολομέλη, αλλά τώρα μιλάμε για τους δημοκρατικούς κανόνες. Και με λυπάμαι, Ντάνη, αλλά δεν είναι δυνατόν έτσι έχουν τα πράγματα, λυπάμαι. Κάνε τι νομίζεις. Δεν είναι προσωπική η επίθεση. Θα πρέπει να είναι σαφές ότι η διάσκεψη των Προέδρων ε, πρέπει να σέβεται τις αρμοδιότητες των επιτροπών. Δεν είναι δυνατόν σε τέτοια θέματα να λειτουργεί έτσι η κατάσταση. όλοι οι πρόεδροι των ομάδων έχουν ευθύνη. Μία απλή παράκληση και να μην υπερβάλλουμε. Να, καθο... να καθίσουμε δηλαδή στην διάσκεψη των Προέδρων και να αναρωτηθούμε γιατί πήγαν τα πράγματα όπως πήγαν. Δεν είναι υπερβολικό αυτό θεωρώ. Δεν είναι υπερβολικό να ζητάμε σεβασμό στις αρμοδιότητες των ε, επιτροπών και ίσω σε κάποια σημεία να υπάρχει ανάγκη να γίνουν διαφορετικά τα πράγματα, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει σε συμφωνία με την Επιτροπή. Συνάδελφε, νομίζω ότι είναι πολύ συμπαθητικά αυτά που είπατε κυρίω για τον ε, κύριο Μπέγκε και νομίζω ότι όλοι συμμεριζόμαστε. Από το Μάιο του 68 έχουμε αυτή την εμπειρία στη Γαλλία. Το να δίνει κανείς την ευκαιρία στο Ντάνι Κομπεντίτ ε, το, το λόγο αναλαμβάνει τον κίνδυνο μετά. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να αντιπαραθέσω οτιδήποτε. Απλά θέλω να πω ότι είμαστε, και αυτό είναι το πρόβλημα στην όλη την παράθεση για τον προπολογισμό, βρισκόμαστε σε μια έντονα πολιτική αντιπαράθεση, η οποία από πλευράς προϋπολογισμού αφενός έχει τη σημασία της, αλλά εκ παραλλήλου έχει και μια σημασία σε ό,τι αφορά την ερμηνεία όσων προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό ε, επεμβαίνει η διάσκεψη των Προεδρών, γιατί στην αντιπαράθεση από τότε που υπάρχει η συνθήκη της Λισαβόνας έχουμε μια αναμέτρηση ισχύω μεταξύ του Συμβουλίου που ερμηνεύει διακυβερνητικά την Λισαβόνα και του Κοινοβουλίου που πράττει διαφορετικά. Επειδή λοιπόν εξ αρχής η κατάσταση η οποία ήταν δύσκολη και για τον Αλάν για παράδειγμα γιατί στην ίδια κατάσταση που χρειάστηκε να διαπραγματευτεί, χρειάστηκε να διαπραγματευτεί και ο Μπούσικ. Το πρόβλημα όμω είναι το εξή, επειδή για πρώτη φορά είναι πολιτική αντιπαράθεση εδώ. Και αυτό υπερβαίνει την αντιπαράθεση για τον προϋπολογισμό. Είναι καθοριστική αντιπαράθεση αυτή μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Και γι' αυτό λοιπόν εξ αρχής υπήρξε αυτή, αυτός ο διχασμός και καταλαβαίνω ότι υπάρχουν προβλήματα, αλλά δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όλοι οι πρόεδροι όλων των ομάδων ανέλαβαν να κάνουν αυτή την αντιπαράθεση. Και για παράδειγμα, επειδή δεν είμαι ικανοποιημένο, επειδή ουσιαστικά μόνο ο Φερχόφστατ και εγώ ε, υποστηρίξαμε τον ε, Λαμασούρ με την ε, σύμβαση, Είχατε λοιπόν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να υποστηρίξετε του προέδρου. Δύο Προέδροι, εγώ και ο Φερχόφστατ, υποστηρίξαμε τον Πρόεδρό σα και όλοι οι υπόλοιποι τον αφήσατε ξεκρέμαστο. Έτσι απλά έχουν τα πράγματα. Μάλλον δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα σε αυτή την παρτίδα, αγαπητέ μου φίλε. Και δυστυχώ θα πρέπει να σηκωθώ να φύγω γιατί έχω υποσχεθεί να κάνω και άλλα πράγματα. Ανά πάσα στιγμή ε, είμαι διατεθειμένος να έρθω και να το συζητήσουμε επί ώρα στο θέμα αυτό με ειδική πρόσκληση. Δεν φεύγω επειδή δεν περνάω καλά. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου. Θα ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που θα σηκωνόμουν να φύγω από μια συζήτηση επειδή απλά ήταν δυσάρεστη για μένα. Θα ήταν υπερβολικά απλό. Καλώ. Σα είχα προειδοποιήσει. Πολλοί ζήτησαν το λόγο, αλλά παρακαλώ να είστε συνοπτικοί γιατί έχουμε και άλλες ψηφοφορίες. Ο κύριος Αρτόγκ. Πρόεδρε, κρίμα που όλοι φεύγουν, ε, γιατί θα θέλω να συζητήσουμε και ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Ποια είναι τα χρήματα τα οποία ε, εξοδεύουμε αυτή τη στιγμή. Ε, είναι νομίζω των κρατών μελών και όχι του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Σα το είχα πει. Θέστε την ερώτηση στον κύριο Κονμπένδιτ. Θα ενθουσιαστεί. Αλλά κατηδίαν παρακαλώ. Γκέραν Φέρμ. Θα είμαι πολύ σύντομο. Σύμφωνα απόλυτα με τον Αλέξανδρ Άλβαρο ότι πρόκειται για μια συζήτηση την οποία θα πρέπει απλά να διεξάγουμε, όχι όμω τώρα. Τώρα, μέσα στην ε, κατάσταση αυτή δεν είναι η κατάλληλη χρονική συγκυρία γιατί υπήρξε όντω μια σύγχυση ω προ τις αρμοδιότητες και οι γραμματείε μπερδεύτηκαν. Μεγάλη σύγχυση επικράτησε. Θα πρέπει αυτό το πρόβλημα να το έχουμε λύσει μέχρι του χρόνου. Αυτό αφενό. Κατά δεύτερον, σε ό,τι αφορά τον Ράιμερ Μπέγκε και το ότι είναι εισηγητή, πραγματικά λυπάμαι για την απόφασή του γιατί θεωρώ ότι ήταν εξαιρετικό εισηγητή. Συμφωνήσαμε μαζί του σχεδόν σε όλα εκτός από το τελευταίο βήμα Κατά τα άλλα, συμφωνήσαμε απόλυτα. Ήταν εξαιρετική η επαφή, συνομιλούσαμε σχεδόν κάθε ημέρα, ήταν εξαιρετικό το έργο τους, πραγματικά λυπάμαι. Και ελπίζω να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση μελλοντικά γιατί είναι το πιο σημαντικό, πιο σημαντική έκθεση πέρα από την έκθεση για τον προπολογισμό και πραγματικά χρειαζόμαστε έναν δυνατό εισηγητή και για το μέλλον. Ευχαριστώ, Γκέραν. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι όλοι εκτιμούμε αυτά που είπατε. Ο Ράιμερ. Ο συνάδελφος Κονπέντιντα έφυγε ήδη, αλλά ήθελα να παρατηρήσω και ίσως η γραμματεία θα μπορούσε να καταρτήσει ένα φάκελο για το πώς ε, η Επιτροπή Προϋπολογισμού εξ αρχής στην ιστορία λοιπόν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάθε χρόνο και κάθε, σε κάθε δημοσιονομική προοπτική χρησιμοποίησε ε, την διαδικασία ε, του προπολογισμού για να κερδίσει πιο πολλά δικαιώματα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αυτή η προσπάθεια της Επιτροπής Προϋπολογισμού την έκανε κάθε φορά μετά το 1979 και σε πολλά βαθμιαία κατάφερε να ε, κερδίσει πιο πολύ δύναμη για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πολύ οι συγητέ το πέτυχαν αυτό στην ιστορία του Κοινοβουλίου και καλό θα ήταν να το υπενθυμίσουμε αυτό για να επανέλθουμε σε μια σωστή και καλή συνεργασία. Merci. Merci. Alors, je vous Ευχαριστούμε. Λοιπόν, προτείνω να περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία στο σημείο 10. Έχουμε τελειώσει τον προπολογισμό. Ερχόμαστε τώρα σε πιο συνηθισμένες εργασίες που νομίζω πιο εύκολα θα βρουν συνένεση ε, μεταφορές. Ο Λάσλο Σούριαν δεν είναι εδώ. Α, ε, εντάξει, μπορούμε να ψηφίσουμε γιατί ο Ζαν Λικντεάν φεύγει. Λοιπόν, έχουμε διάφορες μεταφορές που κατά την άποψή μου μπορούμε, εμβάσματα, τα οποία μπορούμε γρήγορα να εξετάσουμε. 60. 60 ήταν ε, η μεταφορά η οποία θα επέτρεπε την χρηματοδότηση της μπανάνας αλλά δεν υπάρχει νομική βάση. Ωστόσο μου είπαν ότι από νομικής άποψης καλύτερα να το ψηφίσουμε για να το απορρίψουμε. Θα αντικατασταθεί από το 66. Από την 66. Προτείνω λοιπόν να απορρίψουμε την 60. Ποιοι είναι υπέρ της μεταφοράς. Κατά. Ευχαριστώ. Αποχές. Απορρίπτεται. Αντίθετα, σας προτείνω εξ ονόματος του εισηγητή να υιοθετήσουμε την 63, την μεταφορά 63, να ψηφίσουμε μπλοκ καλύτερα για να τελειώνουμε. Αρκετά νομίζω έχουμε παιδευτεί. Λοιπόν, 63, 65 και 66 μεταφορές είναι η συνέχεια μιας πολιτικής συμφωνίας που έγινε στον τριμερή διάλογο όπου κάποια φάση που το Συμβούλιο δέχτηκε να μην ακούει, ότι δηλαδή ελλείψη ελλείψη ε, ε, ε, μάλλον άλλων κονδυλίων μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη γραμμή ICI και τη... για να χρηματοδοτηθεί η μπανάνα και θα βρίσκαμε τον τρόπο για να βάλουμε αυτά τα, αυτά τα χρήματα στα ζεστά, δηλαδή να τα προφυλάξουμε για να χρησιμοποιηθούν του χρόνου για την μπανάνα και το ICI και για να χρησιμοποιηθούν άμεσα για να αντιμετωπιστούν δύο δραματικές επίγουσες καταστάσεις, δραματικές στη Αϊτή και Πακιστάν. Γνωρίζετε την κατάσταση. Αυτή η πολιτική συμφωνία μεταφράζεται σε τρεις μεταφορές, την 63, 65 και 66 και υπάρχει και μια μεταφορά για την καθάριση των γεωρικών λογαριασμών. Δεν είναι πολιτικό θέμα, είναι τεχνικό και τα ψηφίζουμε λοιπόν unblock. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δύο κατά. Αποχές. Εγκρίνονται οι μεταφορές αυτές. Ο Βλαδιμίρ Μάνκα έχει άλλες μεταφορές να μας προτείνει για τα άλλα θεσμικά όργανα. Κύριε Σιγητά, E, e, Πρόεδρε. Τρει ε, μεταφορέ έχω για το SC13 για την αγορά κτηρίων στη Σόφια. Αναβλήθηκε την προηγούμενη φορά γιατί είναι η κυρία Χόλμαϊρ η συγκήτρια. Θα ήθελα να το ψηφίσουμε, αλλά έχω κάποιες ερωτήσεις για το κατά πόσον όλα τα νομικά θέματα που προκύπτουν από τα κτίρια αυτά έχουν ρυθμιστεί. Και ένα δεύτερο ζήτημα αφορά το ότι τα κτίρια αυτά θα εξυπηρετήσουν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά 40% το Κοινοβούλιο, κατά 60% την Επιτροπή. Έχουν ρυθμιστεί όλα τα ε, ποσά και όλε οι ημερομηνίε. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από την εισηγήτρια να πάρει το λόγο και να μα απαντήσει. Ευχαριστώ. Ζήτησε το λόγο ο κύριος Χάρτον και μετά η κυρία Χολμάγερ θα απαντήσει και στους δύο αν είναι ερώτηση. Ο κύριος Χάρτονγκ. Πρόεδρε, να ακούσω τι έχει να πει η συγκητρία πρώτα. Μόνικα, Μόνικα, ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς, ε, είναι πολύ δικαιολογημένο το ερώτημα. Σήμερα θέλουμε να κάνουμε μόνο μία μεταφορά ακριβώς επειδή, όπως ανέφερε ο συνάδελφος, ε, υπάρχουν κάποια νομικά ζητήματα τα οποία δεν έχουν ρυθμιστεί 100%. Θα ήθελα λοιπόν να εξηγήσω και να ζητήσω την υποστήριξή σας σε ό,τι αφορά αυτά που υποστηρίζω έναντι του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Πρόκειται για ένα κέντρο ενημέρωσης. Ε, το κτίριο αυτό έχει στο εσωτερικό του και άλλους ε, ιδιοκτήτες. Έχει μάλλον και άλλους ιδιοκτήτες. Είχα υποστηρίξει ότι οι ιδιοκτήτες θα έπρεπε να συμφωνήσουν σε περίπτωση που ενοικιάσουν κάποιους ορόφους να μην μπορούν να τον νοικιάσουν σε οργανώσεις για παράδειγμα ε, οι οποίες ήταν αμφισβητούμενες ε, ή ενδεχομένως κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην προκύψει κάτι τέτοιο στο κτίριο αυτό έξαφνα. Αν λοιπόν οι συνδιοκτήτες δεν συμφωνήσουν να υποχρεωθούν σε ό,τι αφορά την εκμίσθωση, θα πρέπει να ε, σκεφτούμε μήπως θα πρέπει να βρούμε κάποιο άλλο κτίριο. Η απόφαση για τη μεταφορά θα ληφθεί την επόμενη χρονιά, όταν θα έχουμε στη διάθεσή μας ε, όλα τα στοιχεία αυτά. Euh, Ευχαριστώ, Μόνικα. Ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μιλάμε για 10 εκατομμύρια τα οποία θα δαπανηθούν για το ευρωπαϊκό αυτό κτίριο. Εξακολουθώ να θεωρώ αδιανόητο το γεγονός ότι δίνουμε σε τέτοιες δύσκολες οικονομικές εποχές τέτοια μεγάλα ποσά. Ευχαριστώ, κυρία Χολμαϊρ. Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για τέτοια πράγματα να έχουμε διαβάσει και τα έγγραφα. Δεν ε, ε, κάνουμε ανακαίνιση όπως είπατε. Αγοράζουμε ένα κτίριο και αυτό σημαίνει ότι στο μέλλον δεν θα πληρώσουμε ε, ενίκιο και δεν δίνουμε 10 εκατομμύρια, δίνουμε 9 εκατομμύρια, το οποίο είναι στην παρούσα φάση χαμηλότερο από την πραγματική αξία του κτηρίου. Άρα αυτό τι σημαίνει ότι θα βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση από ό,τι βρισκόμαστε έως τώρα, που πληρώναμε κάθε μήνα υψηλά ενίκια. Άρα η απόφαση του Κοινοβουλίου να αγοράσει και μάλιστα έναντι των σωστών τιμών για να έχουμε και ένα κέρδος, σε αυτή τη βάση εργαζόμαστε και όχι σε οποιαδήποτε άλλη βάση. Ευχαριστώ κύριε Μποκός. Καταρχάς θα ήθελα να ζητήσω με σεβασμό από τον Πρόεδρο να επαναφέρει την τάξη στην αίθουσα. Δεν ακούμε τίποτε. Είναι αδιανόητο, είναι απίστευτο. Ο κύριος Μποκρός έχει δίκιο. Ζητώ από όσους δεν επιθυμούν να συμμετέχουν ή να παρακολουθούν τη συνεδρίαση να εγκαταλείψουν την αίθουσα. Οι υπόλοιποι σιωπή παρακαλώ. Κύριε Μπούκρος. Σας ευχαριστώ. Ένα άλλο σημαντικό θέμα που ήθελα να θέσω. Εξακολουθούμε να μην καταλαβαίνουμε γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρειάζεται κτίρια σε οποιαδήποτε πρωτεύουσα. Δεν είναι θέμα κτηριακής πολιτικής προφανώς, ωστόσο θα καταψηφίσουμε το θέμα αυτό, γιατί δεν βλέπουμε γιατί θα πρέπει να υπάρχουν τέτοια κτίρια. Κύριε Σαρτούγκ. Πρόεδρε, χαίρομαι ιδιαίτερα με την παρατήρηση που έκανε ο συνάδελφος Μπόκρος. Ακόμα και δύο εκατομμύρια να δίνονται. Μια τέτοια πολιτική απόφαση σε αυτή τη δύσκολη στιγμή της κρίσης Ε, γιατί να δίνουμε τέτοια χρήματα για ένα τεράστιο και όμορφο κτίριο στην Σόφια ενώ θα αρκούσε μια αντιπροσωπεία. Είναι πραγματικά απίστευτο το ότι γελάτε, ενώ οι άνθρωποι στην Ιρλανδία πλήττονται τόσο πολύ από την κρίση. Πραγματικά το θεωρώ εξευτελιστικό σχεδόν. Η κυρία Ολμάιερ. Θα είμαι σύντομη και περιεκτική. Το κέντρο ενημέρωσης, το γραφείο ενημέρωσης δεν είναι μόνο του Κοινοβουλίου, αλλά εξυπηρετεί και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή το κάνουμε από κοινό και κατά δεύτερον εξοικονομούμε χρήματα επειδή αγοράζουμε και δεν ενοικιάζουμε πλέον. Σε περίπτωση λοιπόν που θα πουλήσουμε πάλι το κτίριο, αυτό τι σημαίνει ότι θα έχουμε κέρδος και άρα είναι υπεύθυνη η συμπεριφορά μας. Γιατί δεν θα πρέπει να κάνουμε αποταμίευση αυτή τη στιγμή, γιατί στο μέλλον αυτό τι θα σήμαινε, ότι θα είχαμε υψηλά νίκη κάθε μήνα και θα ξοδεύαμε πιο πολλά χρήματα. Επίση, λέτε ότι δεν θέλετε να δίνουμε σε καμία πρωτεύουσα των 27 κρατών μελών ενημέρωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν ανταποκρίνεται σε αυτά που έχει αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλιώ έχουμε αποφασίσει. Έχουμε αποφασίσει να δημιουργήσουμε γραφεία ενημέρωση και να πω και στον κύριο Μάνκα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρηματοδοτήσει πλήρως το 60% το ποσοστό δηλαδή που της αναλογεί. Αυτό το έχουμε αποφασίσει από κοινού με την Επιτροπή. Πολύ ωραία. Τελευταία φορά θα δώσω το λόγο στον κύριο Ποκρό και στον κύριο Χάρτογκ που το ζήτησαν και μετά θα ζητήσω από τον εισηγητή μας να ολοκληρώσει. Ο κύριος Μποκρός, δεν θέλω να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση επαόριστον και προφανώς συμφωνώ με τον Πρόεδρο ότι πρέπει να τελειώσουμε και τις εργασίες μας. Απλά για τα πρακτικά θα ήθελα να πω ότι δεν πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε καμία περίπτωση χρειάζεται χώρο στη Σόφια ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος για αυτά που είπατε ότι είναι, μάλλον σε σχέση με αυτά που είπατε, πρόκειται για μια αποταμίευση. Σε σχέση όμω με αυτά που εννοώ εγώ, δεν πρόκειται για αποταμίευση. Ευχαριστώ, κύριε Σαρτόγκ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Δεν νομίζω ότι μπορώ να πείσω την κυρία Χόλμαϊερ. Αλλά εξακολουθώ να θεωρώ απίστευτο το γεγονός ότι θεωρεί ότι τα 10 εκατομμύρια είναι αποταμίευση. Θα ήθελα απλά να ζητήσω σεβασμό Προ του βουλευτέ οι οποίοι έχουν ε, διαφορετική άποψη από την ίδια την κυρία Χολμάιερ. Καλώς, σεβόμαστε πλήρω όλους τους ευρωβουλευτέ και ρημνώ και προσωπικά γι' αυτό. Δεν ξέρω τι γίνεται στι δικές σας πατρίδες. Πάντως εγώ εκλέγομαι στην Ανατολική Γαλλία και στην ε, Γαλλία λαμβάνονται κεντρικά όλε οι αποφάσει Η κυβέρνηση βρίσκονται στο Παρίσι, αλλά όλες οι επαγγελματικέ οργανώσεις, οι επιχειρήσεις, μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, εδρεύουν στο Παρίσι. Και για να γίνει βάθηση όλων αυτών των φαγγέλων, χρειάζεται να έρθει σε επαφή με όλους τους εκπροσώπους των ενδιαφερομένων στη Γαλλία. Ή κάποιοι ενδιαφερόμενοι έρχονται και με βρίσκουν, ή δημοσιογράφοι μου ζητούν ε, συνέντευξη, αλλά όλοι οι δημοσιογράφοι δουλεύουν στο Παρίσι. Αν δεν υπάρχει γραφείο για να υποδέχεται τους ε, Γάλλους ευρωβουλευτές στο Παρίσι, πού θα δουλέψουν. Τι θα πάω στο καφενείο ή θα πάω στους λομπίστες, στις ομάδες πίεσης. Νομίζω ότι είναι θέμα αξιοπρέπειας κοινοβουλευτικής και σοβαρότητας του έργου μας. Χρειαζόμαστε γραφείο στο, στη Γαλλία, στο Παρίσι, μοιραζόμαστε 29 ευρωβουλευτέ σε ένα γραφείο. Ωραίο γραφείο. Η κυρία Γκρελιέ έχει το δικό της γραφείο στον πάνω όροφο, που επίσης μοιράζεται με άλλους τόσους. Ε, γίνονται και σπατάλες, αλλά δεν νομίζω σε αυτό το τομέα να γίνονται. Για να δούμε τι θα μας προτείνει ο εισηγητής για την ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι το κτίριο αυτό ακολουθεί την μεσοπρόθεσμη στρατηγική για την κτηριακή πολιτική που υιοθετήθηκε το Μάρτιο και είναι πολύ καλύτερη αυτή η λύση από τη μίσθωση. Το θέμα είναι πώς θα διαθετηθούν τα νομικά ζητήματα. Αυτό θα το μάθουμε κατά πάσα πιθανότητα του χρόνου. Να μας πει η Επιτροπή πώς θα πληρώνει και σε τι χρονικό διάστημα θα γίνονται οι πληρωμές, γιατί θα πρέπει και εμάς να μας εξυπηρετεί αυτός ο διακανονισμός. Πάντως, σας ε, προτείνω να υπερψηφίσουμε τη μεταφορά και τα άλλα θέματα θα τα επιλύσουμε άλλη στιγμή. Καλώς. Μία διευκρίνηση και ας με διορθώσει ο εισηγητής αν κάνω λάθος. Μου είπαν ότι για το C13 μάθα, ε, λάβαμε επιστολή με μία τεχνική διόρθωση. Οπότε το ποσό είναι χαμηλότερο. Είναι 9.240.000 και όχι 9.900.000. Εντάξει, τα έξι μεγέθους είναι ίδια. Ποιος είναι υπέρ της μεταφοράς που μας ε, συστήνει ο εισηγητής μας. Ευχαριστώ. Κατά, φαντάζομαι ότι μερικοί είναι κατά. Όντως. Πέντε. Αποχές, ωραία, εγκρίνεται η μεταφορά. Άλλη μεταφορά, κυρία εισηγητά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν από μία εβδομάδα ψηφίσαμε έξι μεταφορές για έξι θεσμικά όργανα. Μια πληρωμή που δεν είχε καταβληθεί για τους μισθούς του 2009 στις 24 ε, Νοεμβρίου ε, βγήκε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και ψηφίσαμε έξι μεταφορές. Δύο έχουμε μπροστά μας λοιπόν σήμερα. Αυτές οι μεταφορές βάσει στατιστικών στοιχείων των κρατών ε, μελών καταρτίστηκαν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περίμενε διαφορετικούς αριθμούς από αυτούς που έλαβε σήμερα. Σήμερα έχουμε μια αύξηση 0,4%. Αυτό σημαίνει μείωση για την ΕΟΚΕ και προτείνω να εγκρίνουμε την πρόταση αυτή. Να ψηφίσουμε, δηλαδή, να υπερψηφίσουμε τη μεταφορά αυτή. Ευχαριστώ. Πρόκειται για τη μεταφορά 3, για την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, έτσι. Ποιος είναι υπέρ. Ευχαριστώ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τελευταία μεταφορά αφορά την Επιτροπή Περιφερειών. 6 για το 2010. 6 του 2010 που συμπληρώνει τη μεταφορά που είχαμε εγκρίνει την περασμένη εβδομάδα, την 5 του 2010. Και αυτή είναι μια προσαρμογή. Και υπακούει στους ίδιους λόγους με την προηγούμενη. Έχω μια ερώτηση προς την Επιτροπή, αν έχουμε κάποιο εκπρόσωπο ή εκπρόσωπο της Επιτροπής Περιφερειών. Η Επιτροπή Περιφερειών κάνει οικονομίες στην εκτύπωση των εγγράφων, για παράδειγμα οι οικονομίες αυτές ελήφθησαν υπόψη στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2011. Πάντως είμαι υπέρ της μεταφοράς. Ω, ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να απαντήσει ως προς τις οικονομίες της Επιτροπής Περιφερειών. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας πω ότι ο υπολογισμός μας ε, στηρίχθηκε σε ενημερωμένα στοιχεία γιατί λάβαμε τα τελευταία στατιστικά στοιχεία πρόσφατα οπότε είχαμε αρχικά για λόγους σύνεση προτείνει το 0,7 που μειώθηκε στο 0,4 που προέκυψε από τα νέα στοιχεία. Η μεταφορά βέβαια 6 δεν αφορά τους μισθούς. Ίσως κόπημα θα ήταν να απαντήσει η ίδια η Επιτροπή Περιφερειών στο θέμα αυτό. Ωραία, αν υπάρχει κάποιος αρμόδιος από την Επιτροπή Περιφερειών για να μας εξηγήσει αυτό το θέμα. Πείτε μας και το όνομά σας αν έχετε την καλοσύνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά τις οικονομίες από την εκτύπωση, αυτό έχει συμπεριληφθεί για τον προϋπολογισμό του 2011. Έχει ληφθεί υπόψη. You are Mr. Είστε ο κύριος Jacobsen. Ο κύριος Jacobsen, ναι. Ωραία, είμαστε ικανοποιημένοι με τις απαντήσεις. Ποιος είναι υπέρ της μεταφοράς κατά αποχές, μία αποχή εγκρίνεται, λέει ο πρόεδρος, δεν έχουμε άλλες μεταφορές. Μας έχει μείνει το τελευταίο θέμα της κτηριακής πολιτικής. και έχουμε την, τον Οργανισμό για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, ΑΣΕΡ. Κυρία Χολμάιερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Η κατάσταση δεν είναι περίπλοκη γιατί το κτίριο το πληρώνει η κυβέρνηση της Σλοβενίας. Αυτό σημαίνει ότι δεν συνεπάγεται αυτό έξοδα για μας αλλά υπάρχει δυνατότητα να συνεχίσει η αξιοποίηση του κτηρίου και γι' αυτό προτείνουμε λοιπόν σήμερα. Αυτό δεν είναι προβληματικό, θα γίνει διαχωνισμός αργότερα και είμαι υπέρ της τοποθέτησης του οργανισμού Acer στο κτίριο αυτό στη Λουμπλιάνα. Καλώς. Οπότε η μας προτείνει να λάβουμε υπόψη αυτό το σχέδιο χωρίς να γνωμοδοτήσουμε όμως. Ποιος είναι υπέρ της θέσης της ηγετρίας. Κατά. Αποχές. Τέσσερις αποχές. Άρα δεν γνωμοδοτούμε. Μιλήσαμε και για το γραφείο της Σόφια. Για το INS. Να πω δύο λόγια. Θα ήθελα σήμερα να είχα καταθέσει μια γνωμοδότηση, αλλά επειδή Μιλάμε για ένα ποσό άνω των 260 εκατομμυρίων ευρώ και πολλά από αυτά τα ποσά δεν έχουν διευκρινιστεί και φαίνεται ότι τα θεσμικά όργανα έχουν πολλά διαφορετικά στοιχεία αντιφατικά για το κτίριο αυτό. Γι' αυτό λοιπόν ζήτησα να οριστούν οριστικά και τελειωτικά. Οι επιφάνειες, οι επιφάνειες που εκμισθώνονται για παράδειγμα. Δεν έχει γίνει αυτό ακόμη και θεωρώ ότι είναι θέμα αρχής και το τονίζω αυτό σήμερα ότι θα πρέπει να συνεχίσει ο προγραμματισμός και είμαι θετική σε ό,τι αφορά το κτίριο αυτό και την εγκατάσταση της υπηρεσίας το γεγονός ότι δεν θέλουμε να γίνει, αυτό να γίνει ψηφοφορία τον Δεκέμβριο δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε υπέρ. Απλά θέλουμε να έχουμε τα σωστά στοιχεία στην διάθεσή μας για να μπορούμε να πάρουμε τη σωστή απόφαση. Ε, Λαμπρά. Όντως, αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Τη στέγαση ε, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Θα σα δώσω το λόγο κυρία Γκρέσλε, μια στιγμούλα. Έχετε την ευκαιρία λοιπόν την περασμένη φορά να μα πείτε κυρία Συγγετρία ότι χρειάζεται περισσότερε πληροφορίε τι οποίε ακόμη περιμένετε βέβαια. Οπότε δεν μπορούμε να λάβουμε απόφαση τώρα, θα περιμένουμε τον Ιανουάριο. Ίγκε Γκρέσλε. Και στι Βρυξέλλε θα απελευθερωθεί ένα κτίριο ε, για πολλά άτομα, 12.000 και θα θέλαμε να ξέρουμε τι θα γίνει με το κτίριο αυτό. Ναι, Πρόεδρε, μία ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα μπορούσε να μας απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά το εξή. Αναφέρθηκε ως τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο 245. Πώς καταλήξαμε Μάλλον πώς καταλήξαμε στην 245 τετραγωνικά μέτρα. Γιατί τα σχετικά στοιχεία είναι εξίσου ασαφή όπως και τα στοιχεία για την επιφάνεια και τα στοιχεία για το προσωπικό. Καλώς. και αυτή η ερώτηση στον κατάλογο των ερωτήσεων που έχουμε θέσει προς την Επιτροπή. Έχω και ένα σχόλιο και νομίζω ότι μετά την ψηφοφορία του προπολογισμού για το επόμενο έτος, καλό θα ήταν επανέλθουμε σε αυτό το θέμα, όταν θα είναι πρόσφορες οι συνθήκες και θα μπορούμε να συζητήσουμε και πιο νυφάλια. Η ίδρυση της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης είχε σχεδιαστεί και είχε αναγγελθεί ως ουδέτερη από δημοσιονομικής άποψη. Έχει ένα μικρό κόστος λειτουργίας που θα επιβαρύνει τον προπολογισμό του 2011, αλλά θα είναι χαμηλό το κόστος αυτό, 3-4 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό που είναι σημαντικό όμως από δημοσιονομική άποψη και είναι κάτι που θα μπορούσε να το πει και ο κύριος Χάρτονγκ για τους φορολογούμενους είναι, τα ίδια άτομα. Είτε επιβάλλεται ο φόρος στην πόλη, είτε στο, στη χώρα, είτε στην Ευρώπη, είτε στον ΟΗΕ, ο φορολογούμενος είναι ο ίδιος από τη στιγμή λοιπόν που ιδρύουμε μια κοινή Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για τις 27 χώρες μέλη, αν προσλάβουμε υπαλλήλους στην Ευρώπη, τους δίνουμε ταξιδιωτικά έξοδα, τους προφέρουμε στέγη, θα πρέπει αντίστοιχα να μειώνεται η συμβολή των κρατών μελών. Γιατί ένας αποσπασμένος υπάλληλο μπορεί να επιβαρύνει τον κοινοτικό προϋπολογισμό, αλλά ελαφρύνει αντίστοιχα τον γαλλικό. Αυτό σημαίνει ουδετερότητα, γενική ουδετερότητα μεταξύ ευρωπαϊκού δηλαδή και εθνικών προϋπολογισμών. Οπότε θα πρέπει να δούμε αυτό που λέμε ενοποίηση των λογαριασμών από λογιστική άποψη. Αυτό τη στιγμή δεν την, έχουμε. Όταν ε, συζητούμε την οικονομική διακυβέρνηση και όταν οι οικονομολόγοι συγκρίνουν τις Ηνωμένε Πολιτείες της Αμερικής με το ευρωπαϊκό σύστημα. Και όταν μιλούμε για το policy mix. Το, λένε το policy mix της ΕΠΑ ΕΕ είναι καταπληκτικό, είναι, καλός, καλ, είναι καλός συντονισμός της δημοσιονομικής πολιτικής που χαράσεται στην Ουάσιγκτον και της νομισματικής που την κάνει η Federal Reserve. Εμείς έχουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως αντίστοιχη της ΦΕΔ, αλλά δεν υπάρχει η αντίστοιχη αρχή για την δημοσιονομική πολιτική. Αλλά έχουμε σημαντικά μέσα οικονομικά που είναι το άθροισμα των ε, εθνικών προϋπολογισμών συν τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Αν θέλουμε λοιπόν ένα μέτρο, ο κύριος Μποκρός βλέπω ενθουσιάστηκε, το συνεπήρε αυτό το θέμα, αν θέλουμε λοιπόν ένα μέτρο για, το οικονομικό, για τον οικονομικό αντίκτυπο των δημοσιονομικών πολιτικών στο σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας που σε μεγάλο βαθμό έχει και ενιαίο νόμισμα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το άθροισμα όλων αυτών των προϋπολογισμών. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να σας αναφέρω την ανησυχία μου. Δεν πρόκειται να ξεκινήσουμε συζήτηση τώρα, θα έχουμε άλλη ευκαιρία να επανέλθουμε. Βέβαια ο κύριος Μπόκρος ζήτησε το λόγο τώρα, θα το δώσω και είναι και το ίδιο. Αλλά προσοχή, γιατί μέχρι στιγμής ο καθένας δούλευε μόνος του, στη γονίτσα του. Και από τη στιγμή που όλα τα κρατημέλη, χωρίς καμία εξαίρεση, μειώνουν τις δαπάνες του, υπάρχει μία πηγή ένα είδος κοίτασμα της οικονομίας που δεν τη σκέφτονται αυτή τη στιγμή. Υπάρχει δυνατότητα εξοδεύοντας 1 ευρώ στις Βρυξέλλες να εξοικονομήσουν 27 ευρώ, 1 ευρώ στο κάθε κράτος μέλος. Και νομίζω ότι αυτό τελικά, αυτό τελικά θέλει η Επιτροπή ΣΟΥΡ, αυτό λέει πρόεδρος και ο συντονιστής στο επιχείρημα για την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Αυτό το νόημα έχει. Καλό είναι λοιπόν να έχουμε μια πιο σφαιρική εικόνα. Τελικά λάθος έκανα γιατί εκεί που ήταν να τελειώσει η συνεδρίαση βλέπω ότι αρχίζει και ανάβει η συζήτηση. Ίγκε. Η δημοσιονομική ουδετερότητα δεν υπάρχει. Αλλά δεν το ξέρουμε αυτό στα σίγουρα, γιατί εδώ υπάρχει μεγάλη αδιαφάνεια. Ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, δώσει 350 εκατομμύρια, το κοινοβούλιο σε 460, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς ε, τίποτε. Ως τώρα δεν έχουμε εκπληρώσει το έργο μας ως υπεύθυνοι για τον προϋπολογισμό. Βλέποντας ε, την ε, σύνθεση του προσωπικού για την εξωτερική ε, για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Και αυτό που πραγματικά βρίσκω πολύ αμφιλεγόμενο είναι το εξής. Αυτή η υπηρεσία είναι το 1 τρίτο από το γερμανικό ε, αντίστοιχο, από την ε, γερμανική αντίστοιχη υπηρεσία. Για το 1 τρίτο όμως του μεγέθους της υπηρεσίας έχουμε 2 τρίτα ε, αντίστοιχους ε, διευθυντές. Είναι πολύ περίεργο λοιπόν αυτό και ούτε είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό. Αυτή η υπηρεσία βασίζεται σε μια ε, ανάπτυξη των ανώτερων θέσεων και αυτό θα πρέπει να το εξηγήσουμε εμείς τον απλό πολίτη και θα ήθελα πάρα πολύ να μου το εξηγήσει κάποιος αυτός, να το ζητήσει κάποιος αυτός που να μην ονομάζεται Γκρέσλε. Στη Γαλλία αυτό αποκαλείται Μεξικάνικο στρατό. Δηλαδή ένα στρατό όπου υπάρχουν περισσότεροι στρατηγοί από ό,τι στρατιώτε. Φαντάρι. <laughs> Είναι αυτό ένα κίνδυνο. Ο κ. Μπόκρο. Χαίρομαι κύριε Πρόεδρε που το θέσατε το θέμα αυτό. But I uh, όμως είναι κάπως παραπλανητικό να συγκρίνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη ΣΥΠΑ. Εύχομαι να το δίκιο. Αλλά να προτείνουμε με κάθε σεβασμό σε πέντε χρόνια να ενισχύσουμε και να πούμε τίποτα άλλο πέρα από τις εξωτερικές ε, υπηρεσίες και να δούμε ότι καμία χώρα δεν θα έβγαζε τίποτα να κάνουμε ενοποίηση και να δούμε ότι καμία, ε, κανένα κράτος μέλος δεν θα, θα εξοικονομούσε τίποτα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιες ε, χώρες, όπως και η Γαλλία, δεν θεωρώ ότι θα αναλάμβανε η Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές από τις εξωτερικές του δράσεις, άρα δεν θεωρώ ότι θα είναι μεγάλη οικονομία. Oui, non mais... Euh, ναι, μα Δυστυχώ. Συμμερίζομαι μαζί σας αυτό το φόβο και γι' αυτό και ανέφερα το θέμα. Βεβαίως, βεβαίως. Έχετε δίκιο, κύριε Άρτογκ. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Ακούγοντα τη συζήτηση αυτή, ανακύπτει και πάλι η συζήτηση του υπερκράτους κατά των καλά και εύρυθμα συνεργαζομένων κρατών μελών. Καταλαβαίνετε ότι είμαι υπέρ των κρατών μελών που καλά συνεργάζονται μεταξύ τους και θεωρώ ότι το EEAS το μόνο που θα συνεπάγεται είναι επιπλέον έξοδα και οι κάτω χώρες δεν έχουν καμία, κανένα συμφέρον να έχουν μια τέτοια υπηρεσία στο βασίλειο του Far Far Away, σε ένα τέτοιο μακρινό μέρος και θα ήθελα να γίνει αναβολή μέχρι το νέο έτος. Γιατί δεν είναι και σαφές κατά πόσον υπάρχει νομική βάση και επαρκής χρηματοδότηση για το EEAS. Euh, λοιπόν, ας σταματήσουμε τώρα αυτή τη συζήτηση, αλλά όπως βλέπετε έχει ζουμί. Λοιπόν, ευχαριστώ τον εισηγητή. Ολοκληρώσαμε και το 12. Τελευταίο σημείο είναι το 13, η επόμενή μας συνεδρίαση, που δεν θα είναι του χρόνου, αλλά θα είναι την επόμενη εβδομάδα. 13 Δεκεμβρίου, 20 και 30, Στρασβούργο, στην αίθουσα ΒΙΚ 100. Ευχαριστώ, λίγα τη συνεδρίαση.